De heer president. Aan hij sturen. Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen allerseits. Ε, επαναλαμβάνεται η Σύνοδο. Καλημέρα σα επίση. Ε, έχουμε την κοινή συζήτηση για την ενέργεια ω πρώτο σημείο στη μέση διατάξη.